Αρχίζουμε την συνεδρίαση. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο 15 που είναι το πρώτο για την απογευματινή μας συνεδρίαση. Σήμερα με τη μερική διάταξη είναι η έκθεση Μικολάσικ. Αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο της πολιτικής για την συνοχή. Και δίνουμε το λόγο στον Μύροσαβ Μικολάσικ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για τα καλά σας λόγια. Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, με μεγάλη μου χαρά ανέλαβα να είμαι συντάκτης για αυτήν την στατική έκθεση του 2010 για την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων 2007-2013. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά έκθεση. Η πρώτη τέτοιου είδους ε, έκθεση επιψηφίστηκε κατά την έκτη κοινοβουλευτική θητεία. Η υλοποίηση και εφαρμογή του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε το τίτλο συνοχή Συνοχής Στρατηγική 2007-2013 για την εφαρμογή των προγραμμάτων 2007-2013». Αυτός ακριβώς ο τίτλος και εκεί έχουμε την πλατφόρμα για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Η πρώτη αυθεντική ανάλυση αυτής της εφαρμογής για τα λειτουργικά προγράμματα επιτέλους είναι δυνατόν να επιτελεστεί. Και πιστεύω προσωπικά ότι οι στρατηγικές εκθέσεις είναι πάρα πολύ αξιόλογες πηγές πληροφοριών για την ενημέρωση της χάραξης πολιτικής γιατί πηγάζουν από τις συστάσεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Επίσης θεωρώ ότι αυτές οι συστάσεις των ε, εκθέσεων αυτών είναι επίσης χρήσιμο υλικό για την προπαρασκευή των εθνικών και ενωσιακών προγραμμάτων πλαισίων. Και άρα θα πρέπει οι άριστες των πρακτικών να υιοθετούνται, να, να, να τυχαίνουμε μίσους και να αποφεύγουμε επίσης τα λάθη του παρελθόντος. Το Κοινοβούλιο θα αναλύσει πώς έκαναν τις επιλογές του το κρατημέλιο όσον αφορά τις ε, προτεραιότητες για τις δαπάνες και ιδίως θα δούμε τις περιφερειακές ανισότητες οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως αρμόζει. Παρ' όλα αυτά, η πραγματική αξία της ε, πολιτικής συνοχής αξιολογείται από τη βάση των αποτελεσμάτων, από τη βάση των επιπτώσεων σε κάθε επίπεδο ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό. Και κατά τη γνώμη μου οι λέξεις κλειδιά, οι φράσεις κλειδιά ίσως είναι οι εξή. Ανάλυση των όσων πρόκειται να ακολουθήσουν, διότι η έκθεση θα συμβάλλει στην προβληματική για το μέλλον της πολιτικής συνοχής στην Ένωση. Τώρα, μία σύντομη εισαγωγή. Θα συντάξω την έκθεση επί τη βάση Τη προναφερθής ανακοίνωση τη Κομισιόν προ το Κοινοβούλιο, Συμβούλιο αλλά και Ελεγκτικό Συνέδριο που ονομάζεται Πολιτική Συνοχή Στρατηγική Έκθεση 2010 για την εφαρμογή των προγραμμάτων 7 έως 13. Δεύτερον, έγγραφο εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο προσάπτεται στην προαναφερθή ανακοίνωση και σε αυτό το έγγραφο εργασία που θα συζητήσουμε σήμερα έχω σταθεί στους σκοπούς του πεδίου εφαρμογής, της έκθεσης εφαρμογής για τον στόχο, την υπόθεση εργασίας, τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αναλύονται στην έκθεση. Επεξεργαζόμενος όλο αυτό το υλικό, ακολούθησα τις προηγούμενες συναφείς εκθέσεις της Επιτροπής μας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβα υπόψη την εθνική νομοθεσία για να μπορέσω να δω πώς τα κρατημέλη κατάλαβαν τις καθημερινές γραμμές σε σχέση με την εφαρμογή του εθνικού πλαισίου αναφοράς και των λειτουργικών προγραμμάτων. Τρίτον, σημασία της έκθεση. Στατηγικέ και λειτουργικά προγράμματα, επιχειρησιακά προγράμματα από τα κράτη-μέλη για την περίοδο 2007-2013. Πρόκειται για την, ε, την πιο αξιόλογη φάση και έχουν γίνει κάποιε ήδη επιλογέ όσον αφορά το επίπεδο εφαρμογή των προγραμμάτων που τυχάνουν συγχρηματοδότηση από τα διορθωτικά ταμεία 7-13. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για δύο λόγου. Πρώτον, έτσι θα έχουμε μία γενική εποπτεία της κατάστασης μετά από 18 μήνες υλοποίησης. Αφού αξιολογήσαμε τις στρατηγικές που συμφωνήσαμε και τους στόχους μας. Επίσης υπάρχει πρακτική αναγκαιότητα να δούμε ποια είναι τα μειονεκτήματα. Πού θα πρέπει να δίνουμε τις προσπαθειές μας και θα πρέπει να αναδείξουμε τις καλύτερες πρακτικές και να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Η χρηματοοικονομική κρίση, η ύφεση, αλλά και οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν για το μέλλον αποδεικνύουν το πόσο σημαντική και σχετική με τη συγκυρία είναι αυτή η έκθεση. Σας τονίζω ότι θα αναλύσουμε την τρέχουσα εφαρμογή αλλά και θα δούμε ποια θα πρέπει να είναι κατάλληλη προσέγγιση για το μέλλον γιατί τώρα κάνουμε ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός και άρα οποιαδήποτε σύσταση για βελτίωση της εφαρμογής κατά αυτή την περίοδο και επίσης θα καλύψουμε και την αρχιτεκτονική της πολιτικής μετά το 2013. Και επομένως ξεκινώ από μία υπόθεση εργασίας. Και λόγω των στοιχείων που υπάρχουν η πολιτική συνοχή αποδεικνύει το πόσο είναι σημαντική γιατί συνέχεια βοηθά την κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον, ε, την οικονομία αλλά όμως υπάρχει ετερογένεια ε, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και αφού ανέλησα πάρα πολλά δεδομένα κατέληξα στο ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες σε πολλές ε, περιπτώσεις για την ε, εφαρμογή και να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις και να υπάρχει μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία, αύξηση των συνεργειών με άλλες πολιτικές της Ένωσης αυτή η δημιουργία των συνεργειών αλλά να μην έχουμε και κατάτμιση των, των πόρων, να έχουμε επίσης έλεγχο και αξιολόγηση των καλύτερων πρακτικών. Τώρα, μεθοδολογία. Προτείνω ένα τέτοιο έγγραφο εργασία που θα συμβάλλει σε επικοδομητικό διάλογο με τα μέλη τη Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη και γι' αυτό θεωρώ ότι όλα τα σημαντικότερα στοιχεία πρόκειται να ληφθούν υπόψη και να αναλυθούν περαιτέρω στην εκθεσή μου, θα σας την υποβάλλω πέρα τις 11 Ιανουαρίου και διμερός. Επίσης πρόκειται να συνεργαστώ, πρόκειται ε, να το κάνω διμερώς ή και πολυμερό, με τους σκιώδεις ηγητές. Αλλά και με οποιονδήποτε άλλον χρειαστεί για αυτή την έκθεση της Επιτροπής μας. Και οι σκιοδησυγητές επίσης, αλλά και εσείς θα μου παράσχετε ό,τι τυχόν πληροφορίες έχετε, τόσο ώστε να τις εντάξω στο κείμενο του σχεδίου της έκθεσης και γι' αυτό παρακαλώ όποιος θέλει από την Επιτροπή μας και όχι μόνο τους σκιοδησυγητές να πούν τις απόψεις τους. Τι πολύτιμε παρατηρήσεις του κατά αυτή την περίοδο, ώστε να εμπλουτίσουμε το σχέδιο του κειμένου με τις ε, επικοδομητικές του ιδέες. Χιούμπνερ, σας ευχαριστούμε για αυτή σα την εισήγηση και πάμε τώρα εις τους σκιώδεις εισηγητές Σρέντερ και τρεμόπουλο. Ελίζαμπεθ Σρέντερ πρώτη. Πρώτα ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε εισηγητά εξηγήσατε την προσέγγισή σας. Δείχνει ότι θα υπάρξει συνεργασία και θα προχωρήσουμε με διαρθρωτικό τρόπο, στο το πω έτσι, στην επεξεργασία της εκθέσεως. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την διαθεσιμότητά σας αυτή. Η έκθεση δυστυχώς δεν είναι μόνο μια αξιολόγηση των στρατηγικών σχεδίων και του τρόπου εφαρμογής τους από τις χώρες μέλη, ταυτόχρονα είναι και μια απόδειξη ότι η διαρθρωτική πολιτική είναι σημαντική πολιτική και δεν μπορεί απλώς να περικοπεί, ούτε μπορεί να διαλυθεί και να μπει σε εκείνα τα περίφημα flagship projects για το 2020. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα να τα πούμε από την αρχή, βλέπω ότι η δομή που προτείνει ο κ. Μικολάσικ τα σέβεται αυτά. Τώρα η εκροή των κονδυλίων πρέπει να αξιολογηθεί και πρέπει και να θεμελιώνεται και στην βάση των έργων που εκτελούνται στις χώρες μέλη, ότι δηλαδή τα χρήματα πάνε κάπου και πιάνουν τόπο και ότι δηλαδή η πολιτική συνοχή πράγματι έχει κάποιο σκοπό, κάποιο νόημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει και κριτική να ασκήσουμε βεβαίως στην χρήση των κονδυλίων αυτών. Έχει σημασία αυτό για την συνοχή της Ευρώπης, για την σημασία των περιφερειών και ούτω καθεξής. Βρίσκω λοιπόν σωστό ότι προβάλλονται οι βέλτιστες πρακτικές αξιολόγησης. Θα ήθελα επίσης, σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση, να κάνω ορισμένα σχόλια Πρώτα για το οικονομικό υπόβαθρο της κρίσης. Είναι σημαντικό μεν αυτό, αλλά εγώ δεν θα το τόνιζα τόσο πολύ. Θα προτιμούσα δηλαδή να ε, χρησιμοποιήσω τον χώρο της εκθέσεως περισσότερο για να αναπτύξω τους στόχους. Η ίδια η κρίση δείχνει ανάγλυφα πόσο σημαντική είναι η στόχη. Υπάρχει και η περίφημη Επιτροπή για την κρίση που θα τα δει αυτά. Δεύτερο, θεωρώ ότι πρέπει να εγκύψουμε πραγματικά στο θέμα της εφαρμογής στις χώρες μέλη και πώς έγινε και η εκροή των χρημάτων και χρήματα που έχουν αφαιρεθεί από την περιφερειακή πολιτική και να εξηγήσουμε ότι θεωρούμε εσφαλμένη την κίνηση αυτή. Εξάλλου, οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν δεν, για αυτές μάλλον, δεν ευθύνονται μοναχά οι περιφέρειες. Ευθύνονται και οι χώρες που είναι καθαροί εισφορείς. Ορισμένες εισφορές καταβλήθηκαν με καθυστέρηση πάνω από έτος. Τα γνωρίζετε κι εσείς αυτά, κυρία ε, Πρόεδρε, ήσασταν τότε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίτροπος. Το τρίτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι ορισμένα σημαντικά του κανονισμού δεν εμφανίζονται τόσο πολύ στην έκθεση όπως θα ήθελα και πράγματα τα οποία είχε περάσει το κοινοβούλιο τότε. Η ρήτρα για την βιωσιμότητα, η ρήτρα για τις εταιρικές σχέσεις καθώς και για την ισότητα των φύλων. Το λεγόμενο gender mainstreaming. Αυτά είναι πράγματα τα που έχουν αποδείξει την αξία τους στην περιφερειακή πολιτική για χρόνια πολλά και που ε, αξιολογούνται πολύ υψηλά στις περιφέρειες. Θα ήθελα λοιπόν να περιληφθούν και αυτά. Πρόκειται για στοιχεία αξιολόγησης της πολιτικής συνοχής που πρέπει να διατηρηθούν. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα σημαντικό μέρος της εκθέσεως θα πρέπει να αφιερωθεί στην πρακτική που χρησιμοποιείται στις αναλύσεις αυτές. Καθώς επίσης να θεμελιώνει για ποιο λόγο θέλουμε να διατηρηθούν τα προαναφερθέντα κριτήρια. Σας ευχαριστώ. Κύριε Τρεμόπουλε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον ε, κύριο Μικολάσικ για την εισήγησή του. Θα ήθελα όμως να προσθέσω κάποια σημεία γιατί κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι κινείται σε πολύ γενικές γραμμές και δεν διαφέρει πολύ από την έκθεση της Επιτροπής. Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια θέματα που αποσιάζουν εντελώς ή κάποια άλλα τα οποία αναφέρονται ελάχιστα. Ε, είμαι της άποψης ότι ο θεσμός του Ευρωκοινοβουλίου, η Επιτροπή μας πρέπει να είναι κριτική σε σχέση με τις εκθέσεις της Επιτροπής και αυτό περιμένουν οι πολίτες που μας έστειλαν εδώ. Η έκθεση αυτή είναι ε, η τρίτη στη σειρά, η πρώτη από την προηγούμενη σας θητεία και η επόμενη από τον κύριο Φαν Νίστερ Λόι. Ε, επομένως, καλά κάνουμε και είμαστε προσεκτικοί Κάνατε λόγο για στρατηγική αναφορά που εισήχθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της προγραμματικής περίοδου. Αναφέρατε τους στόχους, την προτινόμενη δομή καθώς και τη μεθοδολογία. Σίγουρα αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία και ε, θα συμφωνήσουμε. Όμως τα σημεία από τα οποία πρέπει να δώσουμε προσοχή είναι τα εξή τρία. Πρώτον, κονδύλια για θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Πολλοί από εμά θα θέλαμε να δούμε όχι απλά να γίνεται λόγος για τις περιβαλλοντικές πολιτικές, αλλά με όχημα την αηφορία και τις προτάσεις για πράσινες επενδύσεις, θα πρέπει να βρεθεί, να αναζητήσουμε φόρμουλα που θα δώσει προοπτική για την ανάπτυξη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, με ταυτόχρονο όμως σεβασμό στο περιβάλλον. Να αναφέρω τα δύο πρόσφατα ατυχήματα, βιομηχανικά, μεγάλης έκτασης στην Ουγγαρία και πιο πριν στη Ρουμανία. Άρα αυτά αηφορία, οικονομική ευημερία πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Το δεύτερο σημείο αφορά τη διαφάνεια. Εδώ αυτή η Επιτροπή έκανε δεκτή την ε, έκθεσή μου για την ε, διαφάνεια και υπερψηφίστηκε τον ε, Ιούνιο με συντριπτική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκεί έγινε σαφές ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για μεγαλύτερη διαφάνεια είναι αδιαπραγμάτευτες. Επομένως, και εδώ θα μπορούσε να γίνει συγκεκριμένη αναφορά για την προαγωγή της ε, διαφάνειας, τις ε, συμβατότητες στην παροχή των πληροφοριών, την συγκρισιμότητα των στοιχείων και άλλα συναφή. Και ένα τρίτο σημείο είναι η αρχή της συνεργασίας. Για τις εφαρμογές των προγραμμάτων θα ήταν σίγουρο πολύ χρήσιμο να συλλέγαμε πληροφορίες ή να παίρναμε τουλάχιστον υπόψη όχι μόνο από τις επίσημες αρχές, είτε τις εθνικές είτε τις τοπικές, αλλά και σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με άλλες τοπικές, κοινωνικές και οικονομικές ομάδες. Τις περισσότερες φορές έχουν τουλάχιστον ενδιαφέροντα στοιχεία και οπτικές, αλλά και αποκλήσεις από τις επίσημες εκθέσεις και επομένως η συνεργασία γίνεται στην πράξη και όχι κατ' Αυτά τα τρία σημεία και ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μποστινάρου. Στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την συνάδελφό μου κυρία Κάντενπαχ που κολλείεται. Θα μεταφέρω λοιπόν το μήνυμα που έχει να εξηγήσει στην Επιτροπή η οποία Κάντενμπαχ θεωρεί ότι η Κομισιόν αναλύει τις στρατηγικές και την εφαρμογή τους από τις επιμέρους χώρες μέλη και ότι διακυβεύονται πολλά χρήματα. Δηλαδή 35,7% του συνολικού κοινοτικού προϋπολογισμού που θα πάει σε προγράμματα περιφερειακής πολιτικής και πολιτικής συνοχής. Για αυτό είναι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων φορολογουμένων τα χρήματα αυτά να δαπανηθούν με τρόπο διαφανή και να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά προς το κοινό καλό. Συμφωνεί η συναδελφός μου με την δομή που προτείνει ο κύριος Νικολάσικ για την έκθεσή του. Θα ε, χρησιμοποιήσουμε την έκθεση της Κομισιόν για να διδαχθούμε από το παρελθόν και το παρόν και να εντοπίσουμε ελλείψεις στην διαδικασία, καθώς επίσης και Τομεί που χρειάζεται κάποια ενίσχυση. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να τονίσουμε τις καλύτερες πρακτικές και να τις καταστήσουμε γνωστές και σε άλλες χώρες μέλη. Ιδιαίτερα δε την γνώση αυτή πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε για τον σχεδιασμό μας της επόμενης χρηματοδοτικής περίοδου που θα αρχίσει το 2014, χωρίς να λησμονούμε ότι από την στιγμή της ε, υποβολής των εκθέσεων μόνο 18 μήνες έχουν περάσει και εξακολουθούμε να βρισκόμαστε μέσα στην κρίση. Οι επόμενες του 2012 λοιπόν, τέλη του 2012 θα, έχουν, θα περιλαμβάνουν περισσότερα στοιχεία. Κύριε Κάντερμαχ θεωρεί ότι ο εισηγητής θέλει να τονίσει ιδιαίτερα την πρόοδο των νέων χωρών μελών για να μειώσουν τις περιφερειακές ανισότητες. Χαίρεται επίσης για το γεγονός ότι ο εισηγητής προωθεί συνέργειες των πόρων στις ε, περιφερειακές ε, πολιτικές όπως αυτές του κεφαλαίου 6. Και η κυρία Κάντερμπαχ θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξουν περισσότερη, περισσότερη συνεργασία και με τα άλλα ταμεία, το κοινωνικό, το περιφερειακό. Μιλώντας με τις ε, περιφερειές γνωρίζει ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν δυσκολίες στο ξεκίνημα των χρηματοδοτικών περιόδων αλλά σε σχέση με την προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο οι νέοι κανόνες έχουν βελτιωθεί σε πολλά σημεία. Ζητεί λοιπόν ενίσχυση των προσπαθειών αυτών ακόμα περισσότερο για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Σε ό,τι αφορά την βοήθεια προς τις περιφέρειες, χαίρεται που οι περιφέρειες μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν τις ε, ενισχύσεις έγκαιρα διότι αυτό αποδεικνύει ότι μπόρεσαν να ακολουθήσουν μια εύκαμπτη προσέγγιση και θα πρέπει αυτή να συνεχιστεί και στο μέλλον. Συμφωνεί με τον εισηγητή ότι χρειάζεται να καταβληθούν και άλλες προσπάθειες σε ορισμένους τομείς, ιδιαίτερα για την ενίσχυση της απόδοσης της εφαρμογής, να αποφευθούν υπερβολικές καθυστερήσεις, να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία και περισσότερες συνέργειες μεταξύ άλλων τομέων πολιτική με άλλου τομεί πολιτικής μάλλον. Η κυρία Κάντενμπαχ θεωρεί ότι δεν πρέπει να ε, ξεμπροστιάσουμε των εισαγωγικών διάφορες χώρες ή περιφέρειες, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε εκείνες οι οποίες προωθούν σημαντικούς στόχους και συμφωνεί με την προτινόμενη δομή από τον κύριο Μικολάσικ. Αναμένει τώρα η κυρία Κάντενμπαχ να δει πώς θα διαμορφωθεί στην πράξη η έκθεση. Εν τέλει η κυρία με παρακάλεσε να τονίσω ότι αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον την στενή συνεργασία με τον κύριο Μικολάση και εισηγητή και τους άλλους συνεισηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Γιάν Όλμπριχτ. Specyfika polityki spójności europejskiej polega na tym, że e, rozpoczyna się nowy okres programowania. Κοιτάξτε, είναι γεγονός πως ξεκινά μια νέα περίοδος προγραμματισμού αλλά ακόμα δεν έχουμε καταμετρήσει τον αντίκτυπο της προηγούμενης περίοδους, περίοδου. Δηλαδή, επιβάλλουμε μια νέα περίοδο προγραμματισμού Πράγμα που σημαίνει ότι οι εκθέσεις μας αποκτούν τεράστια σημασία, διότι επηρεάζουν το σύστημα εφαρμογής. Είμαστε στο 2010 και ξεκινάει η συζήτηση για την επόμενη, τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Άρα λοιπόν είναι η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε για τις προοπτικές μετά το 2013. Όπως είπα, δεν έχουμε ακόμα ενδεικτικά στοιχεία για τον αντίκτυπο της προηγούμενης περίοδου. Όμως ε, το, η έκθεση αυτή έτσι και δεν έχει σχέση με το σύστημα συλλογής των στοιχείων αλλά με το θέμα της εκτέλεσης. Η προσέγγιση λοιπόν του κυρίου Νικολάσικ είναι πολύ θετική διότι είναι ιδιαίτερα ευρεία και προτείνει προβλήματα για να βγούμε από το ε, προτείνει μάλλον λύσεις για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ε, προκλήθηκαν κατά την περίοδο 2007 με 2013 και για να δούμε κατά πόσο και σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται αυτές οι πολιτικές που προετοιμάζουμε. Πρέπει με τέτοιο τρόπο να ε, προετοιμαστούμε, να δούμε δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες να δούμε δηλαδή αν τα όσα εφαρμόζονται μετά ελέγχονται, αν υπάρχει σύνδεση πραγματική ανάμεσα στα προβλήματα και τους στρατηγικούς δείκτες οι δείκτες αυτοί μας δίνουν πραγματικά λύσεις. Κατά τη διάρκεια της, ε, περίοδου, της τελευταίας περίοδου αλλάξαμε τον κανονισμό, θα πρέπει να θυμηθούμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό ε, οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν το σύστημα εκτέλεσης των προγραμμάτων. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας Δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε για τα μελλοντικά προγράμματα, γιατί ακόμα αξιολογούμε τα προηγούμενα. Είναι όμως η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε το αν θα συνεχιστούν τα προγράμματα της περίοδου 2007 μέχρι 2013. Να δούμε δηλαδή ποια ήταν τα αδύναμα σημεία και ποια τα δυνατά σημεία της προηγούμενης περίοδου. Το υλικό που έχει συγκεντρώσει ο κ. Νικολάσικ είναι πολύ σημαντικό και έτσι θα μπορέσουμε να εστιάσουμε με σωστές βάσεις στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Λαμπέρτ Φαν Ρόι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετική προσέγγιση, συμφωνώ και εγώ. Ίσως θα μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερη προσοχή στις ε, πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις, τα όσα έλεγε δηλαδή ο συνάδελφος Όλμπριχτ, πώς εφαρμόστηκαν όλα αυτά. Αυτή είναι η καρδιά της έκθεσης. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, προσπαθούμε να αποδείξουμε και κάτι, ότι δηλαδή μια οριζόντια πολιτική, αν και ακόμα και αν εστιάσουμε την προσοχή σε ορισμένους τομείς για να ενθαρρύνουμε την οικονομία ή να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση, στις περιφέρειες όλα αυτά ε, γίνονται με οριζόντιο τρόπο και είναι δυνατό να εφαρμοστεί μια τέτοια προσέγγιση. Αυτό το στοιχείο είναι πολύ σημαντικό γιατί φτάνουμε σε μια φάση όπου η περιφερειακή πολιτική συνοχής θα πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκρισμένα εκτελεστικά μέσα της στρατηγικής 2020. Ο κύριος ε, Μποστινάρο, παραθέτοντας την κυρία Κάντενμπαχ είπε ότι επιθυμεί ακριβώς αυτήν την ε, συνέργεια. Αν πραγματικά αυτά τα συνδέσουμε με την οριζόντια προσέγγιση, λειτουργούν όλα αυτά. Στην έκθεσή μου, την οποία μάλιστα παραθέσατε και σας ευχαριστώ γι' αυτό, εγώ έλεγα ότι αυτή η συνέργεια θα πρέπει να αναπτυχθεί σε σημαντικούς ε, τομείς και προς σημαντικές κατευθύνσεις διότι είναι πολύ σημαντική για τα πανεπιστήμια, τις επιχειρήσεις, τους δήμους, όλους τους σημαντικούς φορείς δηλαδή για τις περιφέρειες. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν στην έκθεσή μου ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποιες είναι οι προτάσεις βελτίωσης και αν όλα αυτά αντιστοιχούν με τις πληροφορίες που μας δίνετε εσείς και η Κομισιόν. Να δούμε δηλαδή στην ουσία αν πετύχαμε τους στόχους μας. Είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η έκθεση αυτή δείχνει ότι τα ε, μέσα για τα οποία επιλέξαμε, δηλαδή να βασιστούμε στην οικονομία της γνώσης και ούτω καθεξής, αν λειτουργούν ή αν μεταφράζονται σε νέες μορφές, νέες συμφωνίες με τα κρατημέλη, ε, συμβάσεις που κάνουμε ή ίσως τους όρους που μπορεί να βάλουμε. Είναι αυτό κάτι το οποίο συχνά ακούω και διαβάζω. Να δούμε δηλαδή πώς λειτουργούν και αν λειτουργούν όλα αυτά. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι η περιφερειακή πολιτική και ο στόχος 2 μεταξύ άλλων είναι ήδη πεπερασμένη, ότι δηλαδή στην εποχή της παγκόσμιας, του παγκόσμιου ανταγωνισμού δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο. Εγώ νομίζω αντίθετα πως πρέπει να αποδείξουμε πως ε, ε, προσφέρει στην συνοχή, την οικονομική και την ε, περιφερειακή ε, αντίθετα. Είμαι λοιπόν έτοιμος να τα συζητήσω όλα αυτά μαζί σας. Πρόεδρος, θέλει κάποιος ακόμα να πάρει το λόγο. Όχι. Πριν να ζητήσω από τον κύριο Μικολάση και να σχολιάσει τα δικά μας, τις δικές μας παρεμβάσεις, να αναφέρω κάτι ακόμα. Πιθανότατα θα γνωρίζετε ότι την περασμένη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ένα έγγραφο εργασίας ε, για την συμβολή μάλλον την ανταπόκριση της πολιτικής στην οικονομική κρίση, πράγμα που θα μπορούσε να σας βοηθήσει στην σύνταξη αυτού το σημείο στην έκθεσή σας όταν μιλάτε για την κρίση. Είναι πολύ πρόσφατο υλικό δηλαδή που θα βοηθήσει στη γενική σας αξιολόγηση. Μπορείτε να σχολιάσετε τώρα αν θέλετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αρχίσω με τα δικά σας λόγια Ασφαλώς θα λάβω υπόψη αυτά που μόλις είπατε, γιατί όντως το υλικό αυτό προσφέρει κάποιες σκέψεις για το μέλλον, για το πώς δηλαδή η κρίση επηρεάζει την κατάσταση στην Ευρώπη. Θα ήθελα επίσης να επεκταθώ λίγο, αποτελεί και καθήκον μου άλλωστε, στη βάση του υλικού αυτού και μέσα στο κείμενο μπορούμε να μιλήσουμε και για τις στρατηγικές εκθέσεις για το μέλλον της ε, ε, πολιτικής συνοχής. Και αυτό θα συμβάλλει στη συζήτηση του θέματος. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτές οι στρατηγικές εκθέσεις να ε, συνεχίσουν και για τις μελλοντικέ ε, πτύχες του θέματος. Θα ευχαριστήσω πρώτα όλες και όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την κυρία Σρέντερ για τα ενδιαφέροντα που είπε και τα σημείωσα προσεκτικά. Και με χαρά θα συνεργαστώ μαζί σας καθώς και με τους άλλους συναδέλφους και της δικής σας πολιτικής ομάδος. Ο κύριος Τρεμόπουλος Ασφαλώς και θα είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος απέναντι στα όσα είπατε. Μπορούμε να λάβουμε υπόψη, ασφαλώς, το έργο σας, την εργασία που έχετε κάνει στον τομέα αυτό και ε, να ενσωματώσουμε καλύτερα κάποια από τα θέματα που αναφέρατε. Ε, είμαι ιδιώδης συνομιλητής για σας γιατί είμαι και μέλος και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, άρα έχω ιδιαίτερη ευαισθησία για τα λόγια σας, για όσα έχετε να πείτε σχετικά με τις περιβαλλοντικές πολιτικές και αν έχετε κάποιες συστάσεις που μπορούμε να ενσωματώσουμε είτε στο κείμενο είτε μέσω τροπολογιών με κάποιο θετικό τρόπο. Ε, για σας κύριε Μποστινάρου που εκπροσωπείτε την αγαπητή μου φίλη κυρία Κάντενμπαχ χαίρομαι που εκφράσατε ικανοποίηση της συναδέλφου μου για την προσέγγιση μου. Η ιδέα αυτή να εξετάσω την σύγκληση και τις συνέργειες αυτές μεταξύ του κοινωνικού και του περιφερειακού ταμείου θεωρώ ότι είναι απαραίτητα. Πρέπει να τα εξετάσουμε δηλαδή και από αυτήν την οπτική. Ευχαριστώ επίσης και τον συνάδελφο Όλμπριχτ που είπε σίγουρα τουλάχιστον ένα σημαντικό πράγμα. Νομίζω μάλιστα ότι είχα δίκιο που δεν άρχισα να απαριθμώ, να σας παραθέτω αριθμούς και ποσοστά για το πόσες χώρες, πόσα έργα. Αυτά είναι θέματα που ενδιαφέρουν τους λογιστές. Παρ' όλα αυτά θα λάβω υπόψη ε, κάποια συγκεκριμένα ε, στοιχεία. Το κείμενο πάντως ε, βρίσκεται σε ένα ενδιάμεσο διάστημα. Δεν έχουμε ακόμα βέβαια όλα τα στοιχεία για να συζητήσουμε πλέον τελεσίδικα. Σε ένα-ενάμιση χρόνο θα έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες, πολύ περισσότερα στοιχεία για να μπορούμε να καταλήξουμε συμπεράσματα. Για τον κύριο Βανίστελ Ρόι έχω μιλήσει και παλαιότερα για καινοτομία, για περιφέρειες, για έρευνα που διεξάγεται στις περιφέρειες. Είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος στις ιδέες που εκφράσατε για τα πανεπιστήμια, για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και θα περιληφθούν και αυτά. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους και με χαρά θα συνεργαστώ μαζί σας. Και για σας κυρία Πρόεδρε μπορώ να διαγράψω, να σκιαγραφίσω σύντομα το, το χρονοδιάγραμμα που μου φαίνεται ρεαλιστικό. Έχουμε λοιπόν σήμερα την πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων. Θα κάνω κάθε δυνατή προσπάθεια για να δώσω το σχέδιό μου στην μετάφραση μεταξύ 7 και 11 Ιανουαρίου. Για μένα η 11η Ιανουαρίου είναι πραγματικά η καταληκτική ημερομηνία για την σύνταξη του σχεδίου μου. Θα το υποβάλω στη μετάφραση λοιπόν τότε. Και ίσως μπορούμε στις 26-27 Ιανουαρίου να προβείτε σε μια πρώτη εξέταση του σχεδίου. Η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών θα πρέπει να οριστεί βέβαια αλλά οι τροπολογίε μεταφρασμένε θα πρέπει να είναι στη διάθεσή μα τον Φεβρουάριο του 2011. Θα προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων επ' αυτών και θα τις εγκρίνουμε στην Επιτροπή Ρέτζι στις 28 Φεβρουαρίου. Νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα αυτό και θα προχωρήσουμε βέβαια στην τελική έγκριση μετά. Αυτή είναι η πρόταση που κάνω. Νομίζω ότι είναι αρκετά ταχύ το χρονοδιάγραμμα αυτό, χωρίς να είναι υπερβολικά. Uh, Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Σημειώνουμε την πρόταση χρονοδιαγράμματος. Η επόμενη βέβαια συνεδρίαση που θα γίνει τον Ιανουάριο, όπως είπατε και εσείς, θα είναι επί του σχεδίου σας. Μπορούμε εδώ λοιπόν να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση του 15 και να προχωρήσουμε στο 16. Βίκτορ Μποστινάρου, σχέδιο γνωμοδότησης για την στρατηγική της Ένωσης για το πλέξι, έκθεση που ε, επί της ουσίας συντάσσει η Επιτροπή Εξωτερικών. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ξεκινήσω λέγοντας η περιοχή αυτή είναι μία από τις πιο σημαντικές αν και είναι τμήμα της Ένωσης αφού μπήκαν στην Ένωση η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Ωστόσο, η περιφέρεια αυτή είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και παρακαλώ να θυμάστε ότι έχουμε δύο κράτη-μέλη ε, της Ένωσης, δύο χώρες που τουλάχιστον επισήμως εξέφρασαν την επιθυμία τους είτε να ε, εισχωρήσουν στην Ένωση είτε να έχουν θεσμικές θέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ουκρανία και τη Μολδαβία. την Τουρκία που είναι κράτος ε, προς ε, ένταξη και έχουμε και βέβαια τον μέγα εταίρο τη Ρωσία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να διερωτηθούμε η Ένωση έχει φωνή η Ένωση για αυτό το τομέα κάνει τίποτα για τις εξελίξεις μπορεί από μόνη της να κάνει τα πάντα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Όχι βέβαια. Χρειάζεται να έχει συνεργασία όχι μόνο με τις χώρες της περιοχής, αλλά και σε ευρύτερες εταιρικέ σχέσεις. Θα ξεκινήσω δηλώνοντας ότι δίνω μεγάλη σημασία στη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, ένα τομέα όπου μετά την προσχώρηση των δύο χωρών η διαδικασία ακόμα εξελίσσεται. Πρόκειται για μια περιφέρεια που ε, παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τον παγκόσμιο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από την άποψη των μεταφορών, της ενέργειας, της, του περιβάλλοντος, ρήπανση, βιοπικιλότητα και μην ξεχνάτε ασφάλεια και σταθερότητα που είναι επίσης πολύ σημαντικό ζήτημα για την ΑΦΕΤ που είναι η αρμόδια της ουσίας επιτροπή για την έκθεση αυτή. Η Ευρώπη σίγουρα θα πρέπει να προωθήσει το ρόλο της στην περιοχή και αυτό σε, με εταιρικέ σχέσεις. Και ακριβώς για τον ίδιο λόγο προσδίδω μεγάλη σημασία σε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την Μαύρη Θάλασσα. Είναι σαφές ότι η ανάπτυξη της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας είναι σημαντική όχι μόνο για τις μεμονωμένες χώρες που βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Ήδη προσπάθησαμε να, δώσουμε να δείξουμε τη σημασία που αποδίδουμε στην περιοχή με την ε, οικονομική συνεργασία στον έξινο πόντο. Αλλά έχουμε συνέργεια, αλλά χωρίς την ενέργεια. Και αναφέρομαι και στην μη πολιτική ενέργεια, όχι μόνο όχι μόνο στην ενέργεια που κινεί τους κινητήρες. Το, το πρώτο συστατικό για την αποτελεσματικότητα είναι η εμπλοκή όλων των χωρών της Μαύρης Θάλασσας χωρίς διάκριση μεταξύ των ε, κρατών που ανήκουν στην Ένωση και αυτών που δεν ανήκουν. Και θα πρέπει να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με τις δύο άλλους βασικούς παίκτες στην περιοχή. Ο ένας είναι η η Θράκη και το, η, η Ρωσία με συγχωρείτε και η άλλη, ο άλλος μεγάλος παράγοντας είναι η Τουρκία. Εγώ προσπάθησα να κάνω μια τέτοια επαφή αλλά δυστυχώς με τη Ρωσία αλλά απέτυχε. Η άλλη απόπειρα με τον επικεφαλή της αντιπροσωπείας της Τουρκίας στις Βρυξέλλες ήταν εξαιρετικά καρποφόρα και πρέπει να ομολογήσω ότι οι απόψεις ήταν, ήταν είτε ταυτόσιμες είτε παρόμοιες παραπλήσεις στα περισσότερα ζητήματα, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα θερμικό Όλες οι προσπάθειες με στόχο την ανάπτυξη της περιφέρειας θα πρέπει να είναι συντονισμένες. πράγμα που σημαίνει πως οι διάφοροι φορείς θα πρέπει να εντοπίσουν τις ε, κοινέ προκλήσεις, τους πόρους που υπάρχουν διαθέσιμοι και έπειτα να ενεργήσουν με συντονισμένο και εναρμονισμένο τρόπο. Πιστεύω πως κάποιοι οργανισμοί που μπορούν να βοηθήσουν για την ολοκλήρωση αυτού του στόχου ήδη υπάρχουν και θα σας αναφέρω κάποιους από αυτούς. Υπάρχει ο Οργανισμός της Οικονομικής Συνεργασίας στον Εύξηνο Πόντο, ο ΣΕΠ, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού Παρευξήνης Συνεργασίας, ΠΑΠΣΕΚ και η Επιτροπή για τη Μαύρη Θάλασσα. Και ανέφερα και προηγουμένως την συνέργεια για την ε, Μαύρη Θάλασσα. Πιστεύω πως όλοι είναι της ίδια άποψη ότι δηλαδή η στρατηγική για την ε, περιφέρεια της μαύρη θαλάσσα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει, όπως αναφέρω στην παράγραφο 3 του σχεδίου γνωμοδότησης, να ακολουθήσει λοιπόν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και τη χρήση θεσμοθετημένων αρχών τη πολιτικής της Ένωση για τη συνοχή, διότι στο σχέδιο γνωμοδότησή μου εκφράζω την ε, το, την γνώμη μας για, γενικά για την ανάπτυξη της περιοχής και όχι ε, τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια και τις εξωτερικές υποθέσεις. Η ε, ε, Μαύρη Θάλασσα είναι πολύ σημαντική. μιλάμε για υποδομές μεταφορών και για υποδομές ενεργειακές που κάθε μήνα που περνάει αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία αν θέλετε, έναν αξιοπρεπή βαθμό συντονισμού είναι απαραίτητο όλα τα προγράμματα να τα διαπραγματευτούμε με τις χώρες που βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα, διότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως οι μεταφορές και η ενέργεια θα αναπτυχθούν με στρατηγικό και βιώσιμο τρόπο. Για το ζήτημα αυτό, στην γνωμοδότηση επιστιάζω την προσοχή ιδιαίτερα στα προγράμματα ανάπτυξης των λιμένων και του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Τονίζω επίσης ότι όχι μόνο είναι απαραίτητο να διαπραγματευτούμε τα προγράμματα με τους διάφορους φορείς, αλλά και τα... να τα αξιολογήσουμε. Να δούμε δηλαδή πού ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κόστος όταν σχεδιάζουμε τέτοια προγράμματα. Θέλουμε ανάπτυξη για την περιοχή, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με βιώσιμο τρόπο και όσο γίνεται με πιο φιλικό τρόπο για το περιβάλλον. Τα πρόσφατα γεγονότα στον κόλπο του Μεξικού καθιστούν σαφέ ότι όταν ε, σχεδιάζουμε τις ε, υποδομές ενέργειας θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις συνέπειες ε, των ατυχημάτων και των καταστροφών τέτοιου τύπου. Και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της Μαύρης Θάλασσας από την άποψη της ενέργειας, μην ξεχνάτε το South Stream και πολλά άλλα ρεύματα ή αγωγούς που είναι υποκατασκευή θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπός τους ε, για την περιοχή αυτή που είναι ούτως ή άλλως μια από τις πιο μολυσμένες όσον αφορά τις περιφερειακές θάλασσες της Ένωσης. Σημασία της εξέβρεσης λοιπόν συμφωνίας και του πώς θα, θα βρούμε συμφωνία ε, τη στιγμή του σχεδιασμού. Ας μην ξεχνάμε φίλοι μου πως το 2011 υποτίθεται πως θα ξεκινήσουν οι εργασίες για τον αγωγό South Stream και έχουμε μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες που θα συμμετέχουν, αλλά δεν έχουμε καμιά ευρωπαϊκή στρατηγική για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προγράμματα. Γιατί όπως και στη Βαλτική θάλασσα μας πούνε είναι ένα εντελώ εμπορικό ε, project και θα το εξετάσουμε μόνο από, τον εμπορικό, από την εμπορική σκοπιά και όχι από την σκοπιά της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Το πρόβλημα όμως του περιβάλλοντος δεν είναι, σχετίζεται μόνο με τα ενεργειακά προγράμματα. Η Μαύρη Θάλασσα είναι ήδη πολύ μολυσμένη και αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα το οποίο θίγω στην γνωμοδότησή μου. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά όλους τους μπλεκόμενους στη Μαύρη Θάλασσα και την κοινή λύση που χρειάζεται για να προστατευτεί το περιβάλλον. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό εδώ είναι το πρόβλημά μας να ε, γίνουν όλα αυτά επί τη βάση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Αυτό θα πρέπει να είναι και το κύριο μας μήνυμα όταν θα συζητάμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία, με την Ουκρανία, με τη Μολδαβία, με την Τουρκία. Και αυτή είναι και η πρώτη μου παρατήρηση, ότι δηλαδή <laughs> μέχρι τώρα όλες μας οι συμφωνίες έγιναν κυρίως διμερώς στη Μαύρη Θάλασσα. Ε, εντάξει, είναι αυτό ίσως πιο αποτελεσματικό, πιο ωφέλιμο για να μιλάμε διμερώς για την ενέργεια. Μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν δεσμεύσεις και τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Όμως, πού βρίσκεται η Ευρώπη. Αν θέλουμε μια στρατηγική ευρωπαϊκή για την ε, Μαύρη Θάλασσα, χρειάζεται να έχουμε ευρωπαϊκές απαντήσεις για τα προβλήματα που σχετίζονται με τη στρατηγική αυτή. Σας ευχαριστώ λοιπόν εκ προημίου για τις συμβολές σας, τη συνεισφορά σας. Θα είμαι ανοιχτό σε κάθε συμβολή των συγκεκριμένων συναδέλφων και Βασικά η ευχή μας είναι περισσότερο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη Μαύρη Θάλασσα, πράγμα που είναι ζωτική σημασία αν θέλουμε να είμαστε ένας βασικός ε, παγκόσμιος παίκτη. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για τη θέρμη με την οποία και την προσήλωση με την οποία ασχολείστε με το θέμα. Σας ευχαριστώ. Ο σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Μποστινάρο. Αυτή η στρατηγική θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την... για την ανάπτυξη της πολιτικής για τη Μαύρη Θάλασσα. Ο κύριος Μποστινάρο υπεγράμισε τη σημασία συμμετοχής και εμπλοκής όλων των χωρών της περιοχής, αλλά και των πιστάμενων οργανισμών που αναφέρατε. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να μην επικαλυφθούν οι δραστηριότητες των διαφόρων αυτών οργανισμών στην ε, περιφέρεια αυτή. Βλέπουμε έλλειψη διοικητικής ικανότητες ή έλλειψη χρηματοδότησης, ε, όπου δηλαδή μια αρχική συνέργεια τελικά οδηγεί σε λιγότερη δραστηριότητα ή, εν πάση σε μία ορατότητα αυτών των οργανισμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εν σε μια ορατοτητα αυτων των αναφέρεται, θα πρέπει να παίξει ε, ηγετικό ρόλο στην περιοχή. Κάποια σχόλια τώρα που έχω να κάνω για τη γνωμοδότησή σας. Ε, θα πρέπει να διασφαλιστεί ο συντονισμός όσον αφορά τις θαλάσσιες τις επιχειρήσεις διάσωσης αλλά και έρευνας. Και αυτό το λέω γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν βυθιστεί διάφορα πλοία, μόνο μερικά ναυτικά μίλια στα νυχτά. Ε, είχαμε για παράδειγμα δύο σκάφη, το Χέρα και το Ποσειδόν, που ε, βυθίστηκαν πολύ κοντά στις ακτές. Μαύρη Θάλασσα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εμπορικό κέντρο διαλευση και αυτό δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Προστασία επίση των ακτογραμμών από πιθανέ επιπτώσεις τη διάβρωση. Επιπλέον, γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ιδιαίτερα στην ε, χώρα μου τη Ρουμανία, έχουμε πολύ μεγάλο πολιτιστικό πλούτο και δυστυχώς αυτό δεν είναι και τόσο γνωστό. Μπορούμε λοιπόν να σκεφτούμε και μέτρα για την πρόθεση του τουρισμού και των πολιτιστικών ανταλλαγών στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Από την άποψη τώρα του περιβάλλοντος θα πρέπει να αυξηθούν οι προσπάθειες για αμοιβαία ευθύνη και κοινέ λύσεις ώστε να μπορέσουμε να καθαρίσουμε την ήδη μολυσμένη Μαύρη Θάλασσα. Το περιβάλλον ε, πρέπει να είναι προτεραιότητα των ε, διαφόρων κοινοτήτων που κατοικούν στην ε, περιοχή. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν και μέσω της εξωτερικής υπηρεσίας, της νέας εξωτερικής υπηρεσίας της Ένωσης, αλλά και αυξάνοντας τους πόρους που, με τους οποίους ε, πρικοδοτούνται τα νέα χρηματοδοτικά μέσα. Δεν θέλω τώρα να μπω στα χωράφια της ΑΦΕΤ, αλλά είχαμε διάφορες ε, παγωμένες και λιγότερο παγωμένες ε, συγκρούσεις, όπως στον Βόρειο Κάφκασο, το κίνδυνο Ισλαμικού εξτρεμισμού στην, στον Νότ, Νότιο Κάφκασο, Ναγκόρνο Καραμπάχα και επίσης ε, η διαφορά μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν. Επίσης ο Δούναβης συνδέεται άμεσα με την Μαύρη Θάλασσα. Συζητάμε ταυτόχρονα το μέλλον της ε, Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το Δούναβη. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να συμπεριλάβουμε προγράμματα που σχετίζονται με τη Μαύρη Θάλασσα, όπως ας πούμε στο περιβάλλον, στο τουρισμό και στις υποδομές. Σα ευχαριστώ και πάλι κύριε Μποστινάρο για τη γνωμοδότησή σας και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Θα την παρακολουθήσω γιατί είμαι και στην Επιτροπή ΑΦΕΤ, την αρμόδια επί τη ουσία. και ελπίζω πως δεν θα είναι μόνο στο προς συμφέρον των δύο κρατών μελών που βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά προς το συμφέρον ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ κύριε Στρομόπουλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Μποστινάρου για τη συνδρομή του στο θέμα της ε, Μαύρης Θάλασσας. Κατά τη γνώμη μου κάλυψε ε, πολλά σημαντικά θέματα. Θα ήθελα να προσθέσω κάποιες ε, και κάποιες άλλες παραμέτρους, να μπω και σε κάποιες λεπτομέρειες, σε κάποια σημεία. Το πρώτο σχόλιο είναι σχετικά με τη ρήπανση στη Μαύρη Θάλασσα από ποταμούς όπως ο Δνήπερος, ο Δούναβης, αλλά και τα πετρελαιοφόρα. Ε, κατά μήκο του Δνήπερου ποταμού στην Ουκρανία υπάρχουν ε, μεγάλοι ε, ρηπαντέ, οι μεγαλύτεροι, αλλά και στον Δούναβη υπάρχουν πυρηνικά εργοστάσια. Το Τσέρναβόντα στη Ρουμανία, το Κοσλοντούι στη Βουλγαρία που θα αντικατασταθεί με αυτό το Μπέλενε που και αυτό χρησιμοποιεί τα νερά του Δούναβη. Γενικά, ο Δούναβης στο μακρύ του ταξίδι μεταξύ των διάφορων χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης καταλήγει επιβαρημένος στη Μαύρη Θάλασσα και χρησιμοποιείται και για υδροηλεκτρικούς σταθμούς και δέχεται και γεωργικά και άλλα απόβλητα. Άρα χρειάζεται και μια συνολική αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης. Αυτά τα απόβλητα λοιπόν πέφτουν στη Μαύρη Θάλασσα και από εκεί όμως μέσα από τα στενά του Βοσπόρου καταλήγουν στο Αιγαίο. Ε, το Αιγαίο, ε, να σημειωθεί, παρουσιάζει 7 φορές περισσότερη ραδιενέργεια από ότι το Ιόνιο πέλαγος που χωρίζει την Ελλάδα από την Ιταλία, χωρίς να υπάρχουν πυρηνικά εργοστάσια στην περιοχή. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έρχονται από τη Μαύρη Θάλασσα. Ξεφεύγουν δηλαδή οι επιπτώσεις από την άμεση περιοχή που συζητάμε. Και φυσικά οι ζημιές στο οικοσύστημα, στον τουρισμό ε, μοιράζονται σε διάφορες χώρες. Επειδή λοιπόν υπάρχουν, ε, ε, η ρήπανση δεν γνωρίζει σύνορα, γι' αυτό και χρειάζεται μια διασυνοριακή συνεργασία ε, για μια συνολική και κοινή διαχείριση του περιβάλλοντος. Τα πετρελαιοφόρα που αναφέρθηκε, όπως είναι γνωστό, πολλές φορές αδειάζουν τα σεντινόνερα, ξεπλένουν τα τυχώματα και όπως γνωρίζετε ρηταρίχνουν μαζί στην θάλασσα ε, και καταλαβαίνετε τους κινδύνους αλλά υπάρχουν όπως υπόθηκε και ε, πιθανές επιπτώσεις από μεγάλα περιβαλλοντικά ατυχήματα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η Μαύρη Θάλασσα δεν ελέγχεται επαρκώς. Ε, είναι μια κλειστή θάλασσα, δεν υπάρχουν δηλαδή ρεύματα και γι' αυτό παραμένει μια ρυπασμένη θάλασσα. Δυστυχώς εκεί δεν ισχύει μόνο η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν χώρες όπως η Ρωσία και η Ουκρανία που δεν έχουν και δεν τηρούν την αντίστοιχη, την απαραίτητη νομοθεσία ε, ενάντια στη ρήπανση. Αλλά και χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προβλήματα στην εφαρμογή. Ε, η ρήπανση λοιπόν είναι από τα σημαντικά θέματα και θα πρέπει να υπάρξει κοινή πολιτική πρόληψης, όχι ε, μετά καταστολής. Πρόληψης λοιπόν των πιθανών περιβαλλοντικών ατυχημάτων και από τους αγωγούς ενέργειας ε, στην περιοχή. Ένα άλλο σημείο ε, αφορά τα μικρά έργα, ε, τα people-to-people projects, τα οποία χρηματοδοτούνται από, το Small Project Fund και τα οποία είναι σημαντικά, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες ή συνοριακές περιοχές. Αυτά τα έργα δεν πρέπει να κοπούν, αυτά τα μικρά έργα, να κοπούν, να παραμεριστούν από τα μεγάλα έργα και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ τέλος και στην ανάγκη για καλύτερες υποδομές και συνδέσεις μέσω των ε, διευρωπαϊκών ε, σιδηροδρόμων, των λιμανιών και των πόλεων. Ε, πόλεις όπως η Κωνσταντζα, η σύνδεσή της με τον Βουκουρέστι, η Βάρνα με τη Σόφια. Υπάρχει ανάγκη για καλύτερη συνεργασία των λιμανιών και θα πρέπει να είναι στόχος αυτή η καλύτερη συνεργασία, όπως και οι θαλάσσιες διαδρομές με τις γειτονικές χώρες, χώρες όπως η Ρωσία, η Ουκρανία, η Γεωργία. Και να υπάρχει βεβαίως και ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο και συντονισμός πολιτικών μεταξύ των λιμανιών και των αηφορικών συνδέσμων με την ενδοχώρα. Όλα αυτά σε μια προοπτική βιώσιμης αηφόρου ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τρεμόπουλο. Ο κύριος Στογιάνοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα θα ήθελα να απευθυνθώ στον Έλληνα συναδελφό μου. Δεν ξέρω από πού διαθέτει τις προφορίες που ανέφερε. Αν ξέρει που ακριβώς είναι το Κοσλοντούι, θα ήθελα να το προσκαλέσω να έρθει στη Βουλγαρία μαζί μου, θα επισκεφθούμε τον σταθμό του Κοσλοντούι και έτσι θα μπορέσει ο ίδιος να δει πώς εργάζεται ο σταθμός αυτός. Διότι είπε ότι θεωρεί μάλλον φαίνεται ο ίδιος ο κ. Τρομόπουλος ότι εφόσον υπάρχει ένας πυρηνικός σταθμός αυτομάτως ρηπαίνει. Δεν είναι σωστό κάτι τέτοιο, ούτε μπορεί να λέγεται, διότι μπορεί να προκαλέσει πανικό στο κοινό. Γι' αυτό ε, προτείνω να δείχνει μεγαλύτερη υπευθυνότητα όταν μιλεί και πολύ ευχαρίστω να οργανώσω μια επίσκεψη να έρθει μαζί μου. Διότι αν υπάρξουν βεβαίω, ε, αν υπάρξει ρίβανση και πέσει στο δούναβι, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Τώρα για τον κύριο Ποστινάρου. Δεν γνωρίζω εάν το γνωρίζετε, αλλά τούτη την εβδομάδα μια μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Τουρκίας Έγινε, αλλά απέτυχε. Διότι ο, ο Τούρκος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μίλησε για Νότια και Βόρεια Κύπρο, κάτι που είναι απαράδεκτο. Γνωρίζετε ποια είναι η θέση μας για την Κύπρο. Για τον λόγο αυτό οι ευρωβουλευτές μποϊκοτάρισαν εν τέλει τις συνεδριάσεις της ε, Μεκτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Δεν ξέρω λοιπόν τι συζητήσατε με τον ε, Τούρκο ε, εκπρόσωπο, εγώ θα έλεγα πάντως παραφράζοντας τους ε, αρχαίους Ρωμαίους, τι με ο Τούρκος εντών αφαιρέντες φοβού τους Τούρκους και, φο... και δώρα φέροντας δηλαδή. Μποστινάρου, πολύ ευχαρίστω να πω στον συνάδελφό μου ότι μιλούμε για περιφερειακή πολιτική και μια περιφερειακή ε, οπτική για τον εύξηνο πόντο. Δεν μιλούμε εδώ για τη σύγκρουση μεταξύ του βόρειου και νότιου τμήματος της Κύπρου. Εγώ στην ατζέντα μου δεν είχα θέματα της Κύπρου. Είχα την ευκαιρία και ευχαριστώ την Ταγμάρα πάλι, διότι με βοήθησε στη σύνταξη της εκθέσεως. Καλύτερα λοιπόν να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση που προκαλείται είτε από έλλειψη πληροφόρησης είτε από έλλειψη κατανόησης. Εδώ είμαστε Επιτροπή περιφερικής ανάπτυξης. Δεν είμαστε κανένα διεθνές δικαστήριο. Απλώς μια προειδοποίηση ήταν αυτή, λέει ο κ. Στογιάννοφ. Κύριοι, δεν πρόκειται να γίνει συζήτηση αυτή τώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, περιοριστούμε σε αυτά που συζητούμε σήμερα. Να συζητήσουμε λοιπόν τώρα την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Προτείνω λοιπόν την 9η Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα, κάτι που θα μας επιτρέψει να ψηφίσουμε στις 30 Νοεμβρίου, διότι φαίνεται ότι η ΑΦΕΤ θα ψηφίσει αρχές Δεκεμβρίου, η Επιτροπή Εξωτερικών δηλαδή. Ενθαρρύνω λοιπόν όλους και όλους να συνεργαστείτε στενά με τον Βίκτορα Μποστινάρου επαναλαμβάνω, 9 Νοεμβρίου, 6 το απόγευμα, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Εκτός αν έχετε κάτι να πείτε ακόμη. Μποστινάρο. Θα μιλήσω για σοβαρά πράγματα τώρα. Θα σχολιάσω τις παρεμβάσεις. Ευχαριστώ πρώτα τον κύριο Κοβάτσεκ. Συμφωνώ με όλα όσα είπε. Και έχω την ίδια γνώμη. Μόνο οι περιορισμοί της εκθέσεως δεν με αφήνουν να διευρυνθώ περισσότερο. Αλλά σίγουρα με την συμβολή σας η έκθεσή μας θα φωτίσει τα προβλήματα που αναφέρατε, όπως για παράδειγμα οι επιχειρήσεις θαλάσσιας έρευνας και σωτηρίας, διασώσεως δηλαδή και ούτω καθεξής. Τώρα, για τη σχέση μεταξύ της στρατηγικής του Δούναβη και της Μαύρης Θάλασσας, αυτό είναι απαραίτητο εγχείρημα. Να αναπτύξουμε δηλαδή στρατηγικά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάνουν άλλοι παγκόσμιοι παίκτες. Απευθύνομαι τώρα στον κύριο Τρεμόπουλο. Ε, συμφωνώ μαζί σας, είναι ε, θάλασσα με βαριά ρήπανση. με ιδιαίτερη σύνθεση των νερών. Κάτω από τα 180 μέτρα βάθος, η συγκέντρωση πολύ τοξικών ουσιών είναι στην ουσία θανάσιμη, που σημαίνει ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο να ε, αντιδράσει κανείς όταν συμβαίνουν καταστροφές στην Μαύρη Θάλασσα. Σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική διάσταση θα προσθέσω ότι ήδη υπάρχει η συνθήκη του Βουκουρεστίου για το περιβάλλον που αποτελεί τμήμα της περιφερειακής συνεργασίας. Το πρόβλημα δεν είναι να υπάρχουν αυτά στα χαρτιά. Γυρίζει πίσω, δεν τον ακούμε καλά. Δεν μιλήσει στο μικρόφωνο του. Θα, αν ζητήσετε τη γνώμη μου πάντως, εγώ θα είμαι υπέρ του να ξεκινήσει με την διαμεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια περιφερειακή συνεργασία για περιβαλλοντικά θέματα, ένας περιφερειακός μηχανισμός δηλαδή, για να ασχολείται με όλα τα περιβαλλοντικά θέματα. Και γιατί να μην συζητήσουμε με τη Ρωσία και με άλλες χώρες, για να υπογράψουμε αλλά και να κυρώσουμε την σύμβαση ΕΣΠΟ πριν ενδεχομένως να προσχωρήσουν οι χώρες αυτές ή τέλος πάντων μέσα στις σχέσεις που έχουμε με τις ε, χώρες αυτές. Γιατί μας λένε ξανά και ξανά ότι η Ρωσία έχει υπογράψει την ΕΣΠΟ. Ναι, όντως την υπέγραψε, αλλά δεν την κύρωσε ποτέ μέχρι τώρα. Γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην προωθήσει το μέγα αυτό έργο. Τέλος. Είναι σημαντικό να υπάρχουν κοινά κοινέ περιφερειακές προδιαγραφέ, σίγουρα σύντομα θα έχουμε τον αγωγό South Stream, να έχουμε λοιπόν κοινέ προδιαγραφέ για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών έργων εκεί. Είμαστε μικρέ χώρε οι οποίε βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλε χώρε, μεγάλου παίκτε, σαν αυτού που ανακατεύονται στην South Stream, είτε πρόκειται για την Gazprom, είτε για την Aeon ή για άλλες παρόμοιες μεγάλες επιχειρήσεις. Όπω μου είπε ένα διπλωμάτη, ωραία είναι αυτά που λέτε για περιφερειακές λύσει, αλλά από όσο ξέρω υπάρχει ένα σημαντικό Πρωθυπουργό Ευρωπαϊκή χώρα που έχει πολύ στενέ σχέσει με έναν μη Ευρωπαίο Πρωθυπουργό και που οι δύο έχουν αποφασίσει να προωθήσουν ταχύτατα το South Stream. Πρόκειται λοιπόν για ε, εξαιρετικά ευρωπαϊκό θέμα. Είναι σωστό αυτό που λέτε λοιπόν κύριε Τριμόπουλε. Ευχαριστώ λοιπόν για τις ε, παρεμβάσεις σας. Θα λάβω υπόψη μου κάθε τροπολογία που θα υποβάλλεται. Τελευταία έκθεση, γνωμοδότηση του Βανίστελ Ρόι για την απόφαση Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για, για το έτος της ενεργούς γύρανσης. Δεν υπάρχει βιασύνη ιδιαίτερη εδώ, αλλά μπορούμε να προβούμε σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Λαμπέρ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Το θέμα είναι λιγότερο πολιτικής σημασίας από ότι το προηγούμενο. Αλλά ο αντίκτυπος στην κοινωνία είναι το ίδιο σημαντικός. Η Ευρώπη ζει μια δημογραφική μετάβαση. Περνάμε από μια σχετικά νέα Ευρώπη σε μια κατάσταση που θα έχουμε λιγότερους εργαζόμενους και περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι άνω το 50, 55, 60 και 80 ακόμη ετών. Διαπιστώνουμε λοιπόν την κατανομή του πληθυσμού στον κόσμο, πώς αυτή μεταβάλλεται. Έχουμε περάσει το 14% στο 7%, θα περάσουμε στο 5% του παγκόσμιου πληθυσμού, όσον αφορά τη γεννητικότητα, πρέπει κανείς να διερωτηθεί τι συμβαίνει. Γι' αυτό και φτιάξαμε αυτό το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γύρανσης. Ο τίτλος υποδεικνύει ότι θα πρέπει να αναλάβουμε κάποια πρωτοβουλία. Θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση που θα σκεφτεί όχι μόνο τους ε, ηλικιωμένους, αλλά και τις σχέσεις ανάμεσα στις γενναίες. Λιγότεροι νέοι και γύρανση. Δύο πράγματα. Η πρόταση αυτή είναι μια νομοθετική πρόταση η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή είναι η Επιτροπή Επασχόλησης και έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις ιδέες μας. Όπως έλεγε και ο προηγούμενος ομιλητής, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις περιφερειακές πτυχές, δηλαδή θα πρέπει να σκεφτούμε τι αγγίζει άμεσα τους ε, ανθρώπους, τι μπορούμε να κάνουμε στις πόλεις, περιφέρειες. Να έχουμε δηλαδή αυτή την οριζόντια προσέγγιση, απασχόληση, συμμετοχή, ε, στέγαση, φροντίδα. Ένα έτος λοιπόν για να συνειδητοποιηθεί το πρόβλημα. Φυσικά δεν είναι κάτι το νέο. Υπάρχουν ολόκληρε περιφέρειες της Ένωσης που ήδη έχουν κάνει αυτή τη μετάβαση. Εγώ συμμετείχα σε μία συνεδρίαση πριν από λίγο καιρό στο Λιμβούργο που ήδη έχει διαπιστωθεί η μείωση του πληθυσμού κατά 27%. Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα στην Επιτροπή την Περιφερειακή. Να τονίσουμε τις περιφερειακές πτυχές, αλλά υπάρχει και η καινοτομία που είναι σημαντική κατά την άποψή μου, δηλαδή οι υπηρεσίες, η ηλεκτρονική υγεία κτλ. Ε, λοιπόν, τι έχουμε προβλέψει. Να μην μακρηγορώ έχω ήδη προετοιμάσει κάποιες τροπολογίες. Θα πρέπει να δώσουμε την γνωμοδότησή μας σε συνεδρίαση το τέλους Νοεμβρίου, αρχών Δεκεμβρίου. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η εβδομάδα 49 και 50, ψηφοφορία 26 και 27 Ιανουαρίου εδώ στην Επιτροπή και έτσι θα ψηφίσουμε, θα, έχουμε μάλλον ε, γκρίνει εγκαίρος για τη ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης που θα γίνει την 1η Φεβρουαρίου. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας και θα λάβω υπόψη τις παρατηρήσεις σας στην έκθεσή μου. Είναι κάποιος έτοιμος να σχολιάσει σήμερα? Μάλιστα, κύριε Στογιανόφ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Είναι μια ξέπαινη πρωτοβουλία αυτή και το λέω αυτό γιατί εγώ είμαι ένας από τους νεότερους ευρωβουλευτές αλλά παρότι αφορά τους ε, πιο ηλικιωμένους στη Βουλγαρία αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα και έχω αναφέρει ότι ανάμεσα στην προηγούμενη θητεία και τη, σημερι... και τη τωρινή η μέση σύνταξη αγαπητοί συνάδελφοι είναι κάτω από τα 100 ευρώ μηνιαίως. Πώς μπορεί ένας ηλικιωμένος πολίτης να ζήσει με τέτοια σύνταξη. Να πληρώσει φάρμακα, να πληρώσει τα βασικά είδη διατροφής. Οι Βούλγαροι συνταξιούχοι είναι θύματα μιας πολιτικής απροθυμίας για επίλυση του προβλήματος. Τώρα η νέα βουλγαρική κυβέρνηση αρχίζει να εισάγει κάποιες μεταρρυθμίσεις και επειδή τώρα βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια της συζήτησης, θα ήθελα να συμπεριληφθεί αυτό στη γνωμοδότηση, ότι δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει μια δραστήρια ζωή για τους συνταξιούχους αν δεν βελτιωθούν τα στάνταρ διαβίωσής τους. Μόνο αν βελτιωθούν οι ευκαιρίες για μια καλύτερη ζωή, για περισσότερη ευημερία θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για, μια τέτοιο, για ένα τέτοιο ε, ευρωπαϊκό έτος ενεργού γύρανσης. Σε άλλες χώρες όπως τη Γερμανία ή την Ιταλία οι συνταξιούχοι δεν αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα. Στη Βουλγαρία όμως χρειάζεται να το αναφέρουμε γιατί διαφορετικά πραγματικά θα είναι τρελό να λέμε στους ανθρώπους ότι αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γύρανσης και πρέπει να το γιορτάζετε. Κέλλη. To uh, Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την έκθεση πρωτοβουλία και είναι κάπως ηρωνία ότι η Επιτροπή μας και η Επιτροπή Απασχόληση μιλούν για κάποιους που βρίσκουν δουλειά, ενώ σε αυτήν την ηλικία συνήθω κανεί παίρνει σύνταξη. Επομένω, θα πρέπει πρώτα-πρώτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουμε κάτι για αυτό που είδαμε τελευταίε εβδομάδε σε Ελλάδα, σε Γαλλία και αλλού, ένταση. Γιατί ακριβώ θέλουν να ανεβάσουν το όριο δεξιοδότηση, το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό. Πρώτα-πρώτα λόγω κόστου οικονομικού και δεύτερον διότι επειδή ευτυχώ ο κόσμο τώρα είναι υγιέστερος Νομίζω ότι θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε ενιαίο όρο συνταξιοδότηση παντού στην Ευρώπη. Και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο κοινή συμφωνία και όχι κάθε χώρα μεμονωμένα να μεταβάλει το καθεστώ. Μερικοί όμω έχουν υπερβολικά χαμηλό. Ξέρω ότι είναι θέμα επικουρικότητα, αλλά θα πρέπει κάποια κατευθυντήρια να δοθεί Νομίζω αυτό θα βοηθούσε. Δεύτερον, έχουμε επίσης το τεράστιο κόστος της ε, συνταξιοδότησης και βέβαια η τομέα της υγείας, όμως έχει γίνει μια σωστή επισήμανση να γίνει ευκολότερο το να ταξιδεύουν συνταξιούχοι και έτσι να δοθεί ε, μια όθηση στον ε, τουρισμό. Να δοθούν γενικά ευκαιρίες με αφορμή της αξιοδότηση. Όμως θα πρέπει να γίνει μια σωστή συζήτηση και έτσι να καταλήξουμε σε κάποιες συστάσεις. Και έτσι όλος ο κόσμος θα έχει κάποια, κάποιο μπούσουλα που θα βαδίσει. Μάν, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Μάνερ, να ευχαριστήσουμε για αυτή την έκθεση, γιατί το θέμα είναι όχι μόνο επίγειο, είναι καυτό και επομένω είναι πάρα πολύ σωστό το ότι τώρα το συζητάμε με τόσο ζωντανό τρόπο στην Επιτροπή μας. Σχεδόν παντού έχει τεθεί το ζήτημα του πώς θα καλυφθούν οι γυριότεροι, τι θα γίνει με τις συντάξεις και εμείς πάντως σαν Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής θα πρέπει να κινηθούμε στα πλαίσια της εντολής μας. Τι θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια της επικουρικότητας, τι πρέπει να γίνει πανευρωπαϊκά, τι θα πρέπει να γίνει για την ανάπτυξη των περιφερειών και να δούμε τι ισχύει σε κάθε περιφέρεια στην Ευρώπη, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία και ετερογένεια. Είναι και θέματα ανταγωνιστικότητας, αν και κυρίως το θέμα είναι περισσότερο ανθρώπινο, περισσότερο κοινωνικό. Όμως και τα οικονομικά έχουν τη σημασία τους και η ανταγωνιστικότητα. Γιατί έχουμε μεγάλες διαφοροποίησεις στις περιφέρειες της Ευρώπης, επομένως είναι σημαντικό να αναζητήσουμε τις άρεστες πρακτικές. Σωστό είναι αυτό που λέει έκθεση ότι σε μερικά σημεία, σε μερικές περιφέρειες έχει αντιμετωπιστεί με επιτυχία το πρόγραμμα. Έχουν βρεθεί κάποιες φόρμουλες για την γύρενση του πληθυσμού. Και έτσι να εξετάσουν πρώτα πρώτα και πού το πρόβλημα της διεθνής του πληθυσμού θα έρθει πρώτα και πού αργότερα. Ε, ευχαριστώ. Ε, κύριε Φανίστεζο, θέλετε να πείτε κάτι. Ναι. Θα λάβω υπόψη τα όσα άκουσα. Και θα πρέπει βέβαια να δούμε το θέμα των επιμέρους περιφερειών της Ένωσης. Θα πρέπει να γίνει ίσως για τις συντάξεις μια χωριστή έκθεση. Δεν λέω ότι θα πρέπει εγώ να πιάσω τη λέξη στο στόμα μου, όμως, όμως, είναι τελικά θέμα κρατών μελών. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα κάνουμε ό,τι κάνουμε για να ενθαρρύνουμε τον κόσμο για τις επόμενες δεκαετίες, για να ζητηθούν κάποιες λύσεις για το μέλλον. Εγώ προσπαθώ να είμαι θετικός και επικεντρώνομαι στις εκδηλώσεις που έχουν καθοριστεί για φέτος. Ένα πράγμα είναι αρμόδιο των Ολυμπιτροπών και άλλο τον είναι κανένα θετικός. Ευχαριστώ, Λάμπερτ. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το σχέδιο του κειμένου θα το έχουμε προσυζήτηση για τη συνάντησή μας κατά τα τέλη Νοεμβρίου. Α, και τώρα συνάδελφοι έχουμε ολοκληρώσει, το έχουμε να συζητήσουμε, δεν ξέρω αν έχουμε τίποτε ε, διάφορα. Και θα έχουμε μια μισή μέρα συνεδρίασης όπως είχαμε τώρα και την επόμενη φορά, τον Νοέμβριο. Ίσως έχουμε και κάποια έκτακτη συνεδρίαση με τον Επίτροπο Χαν. σε σχέση με κάποια έκθεση. Οπότε ίσω ε, να τα συζητήσουμε και σε συνάντηση συντονιστών. Η οποία θα ανοιχτεί σε όλου. Γιατί ίσω έχουμε έκτακτη συνάντηση. Έκτακτη συνάντηση και θα το μάθετε τελευταία στιγμή. Αλλά και τον Δεκέμβριο στην τακτή ημερομηνία μας θα τα πούμε και θα γίνει ανταλλαγή απόψεων μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Επομένω, όλοι εδώ ολοκληρώσαμε τι εργασίε μα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ όσου έμειναν στη συνεδρίαση. Γεια σας.